Μία ανακοίνωση. Σας παρακαλώ λοιπόν να με προσέξετε. Χθες ο Πρόεδρος ανακοίνωσε δύο ερμηνείες κανόνων του άρθρου 130 παράγραφος 3 και του άρθρου 191 που προτάθηκαν από την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 226, επειδή δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις προς αυτές τις ερμηνείες, θεωρείται ότι αυτές οι ερμηνείες ενεκρίθησαν. Αυτή ήταν η ανακοίνωσή μου.